ενημέρωσαν για την ε, απόφαση του δικαστηρίου της περιφέρειας της Γκρίμα για μια ποινική διαδικασία κατά του κυρίου Βίνκλερ κατά την άρση της του, μετά την άρση της ασυλίας του, ε, βάσει αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 12 Απριλίου του 2016. Στις 12 ε, Απριλίου του 2018 η διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε